των τροφίμων διαβίβασε διόρθωση σε κείμενο που είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του κανονισμού, η εν λόγω διόρθωση θεωρείται εγκριθήσα, εκτός εάν εντός 24 ωρών από την ανακοίνωση μια πολιτική ομάδα ή ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός ευρωβουλευτών ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία. Το τροποποιητικό κείμενο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Ολομέλειας και ο τίτλος του θα δημοσιευτεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.